Dear και αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε θέμα υπαριθμών 5 της ημερησίας διατάξεως, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Πομιανόφσκι του European Endowment for Democracy. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών, καλώς ήρθατε σήμερα. Η κίνησή σας, Ευρωπαϊκή Στήριξη για την Δημοκρατία, παρουσιάζει την ετήσια εκθεσή ε, από το 2013 δραστηριοποιείστε ε, και έχετε ε, κάνει σημαντικές ενέργειες και προσπάθειες για οργανώσεις που στηρίζουν τη δημοκρατία. Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της. Παρ' όλα αυτά είστε ανεξάρτητη οργάνωση και η προστιθέμενη αξία που προσφέρετε είναι η ευκαμψία που σας επιτρέπει να προσφέρετε ταχεία χρηματοδότηση μέσα σε δύο ημέρες μάλιστα, μέχρι και δύο ημέρες, για οργανώσεις που έχουν ε, δυσκολία εξασφάλισης χρηματοδοτήσεως. Έχετε ήδη μέχρι τώρα χρηματοδοτήσει 250 πρωτοβουλίες και από την αρχή του, 200, του, 2015 ε, έχετε ε, προβεί σε χρηματοδοτήσεις και τώρα μάλιστα χρηματοδοτείτε το πρόγραμμα ε, Γείτονε υπέρ των γειτόνων. Και θα σας δώσω τώρα μέσα το λόγο για να κάνετε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε για την πρόσκλησή σας. Είναι πραγματική, ε, πραγματικό προνόμιο που βρισκόμαστε εδώ και αποτελεί επιβεβαίωση της στήριξης του Κοινοβουλίου προς την εργασία μας. Διορθώνω έναν αριθμό. 400 project έχουμε χρηματοδοτήσει από την αρχή της δραστηριότητάς μας το 2013 και όχι μόνο 250 όπως είπατε εσείς. Μεγάλη ευκαιρία αυτή για μας και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που με έχετε προσκαλέσει και έχω τη δυνατότητα να σας υποβάλω την ετήσια εκθεσή μας, την οποία σας έχουμε διανύμει. Σας δείχνω εδώ το τεύχος είναι φρεσκοτυπωμένη της η έκθεση για το 2016 και μάλιστα υπάρχει διαθέσιμη και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα μας. Προσφέρει πολλές λεπτομέρειες που δεν έχω βεβαίως τον χρόνο να σας εξηγήσω στη διάρκεια της σύντομης παρουσίασης και θα σας παρακαλέσω να δείξετε υπομονή και να διαβάσετε το φυλάδιό μας αυτό ε, διαδικτυακά, αν θέλετε. Το 2016 δεν ήταν εύκολη χρονιά για τη δημοκρατία και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε, τα πάντα άλλαξαν και έγιναν πολύ εντονότερες οι προκλήσεις, παρόλο που προσφέρουμε και νέες δυνατότητες, ταυτόχρονα και ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα πολιτάρχικα καθεστώτα γίνονται ε, χειρότερα σε μια προσπάθεια να φημώσουν τον ελεύθερο λόγο και θυμίζω μόνο την Αίγυπτο, τη Ρωσία και το Αζερβαϊτζάν μάλιστα και πολύ εξελιγμένες ε, εκστρατείες παραπληροφόρησης προσπαθούν να παραπλανήσουν. Θα είδατε το 2016 εξάλλου ότι ορισμένες κυβερνήσεις στην άμεση γειτονία έχουν προσπαθήσει να επηρεάσουν το έργο μας και των εταίρων μας. Δείχνει αυτό βέβαια ότι το έργο μας έχει κάποια απόδοση. Ταυτόχρονα ήταν πολύ σημαντικό που διαθέτουμε κατανόηση και υποστήριξη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ ταυτοχρόνως παραμένουμε απολύτως αυτόνομοι σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτικές μας αποφάσεις. Το 2016 συνεχίστηκε η διεύρυνση της γεωγραφικής μας εντολής, υποστηρίζουμε και τους γείτονες των γειτόνων πλέον, εκτός δηλαδή από τις χώρες της ε, ευρωπαϊκής γειτονίας. Στο πλαίσιο αυτό βασιζόμαστε επίσης στην εισφορά των ευρωπαϊκών θεσμών. Πρόσφατα συναντήθηκα με τον πρέσβη κ. Γκούριαν, ειδικό απεσταλμένο για τις ε, χώρες κεντρικής Ευρώπης και συγγνώμη, της κεντρικής Ασίας για να ε, συζητήσουμε τη στρατηγική του για την Κεντρική Ασία. Σύντομη επισκόπηση των πιο βασικών σημείων της εργασίας μας του 2016 και μετά να σας θέσω υπόψη και κάποιους προβληματισμούς για τη συνοχιζόμενη εργασία μας και τα ζητήματα soft power, τα οποία γίνονται όλο και περισσότερο τμήματα hard security issues. Συνεχίσαμε λοιπόν την ενίσχυση της ε, συνεργασίας μας ως EED. Μέσα στο 2016 διαθέσαμε περίπου 10 εκατομμύρια ε, ευρώ για να ενισχύσουμε 180 έργα, προσπάθειες. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ακτιβιστές την ύπαρξή μας και να αντιλαμβάνονται πώς μπορούμε να στηρίξουμε. Το ίδιο είναι σημαντικό η κατανόηση για το έργο της EED που είναι τα αρχικά μας και στις Βρυξέλλες και στις άλλες πρωτεύουσε, διότι ο ρόλος μας είναι συμπληρωματικό των έργων που αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις. Και χρειάζεται βεβαίω και η πολιτική στήριξη και η ελευθερία δραστηριότητάς μας, για να μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς ε, τα εργαδία μας. 21 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο Διοικητικό μας Συμβούλιο συμμετέχουν στη χρηματοδότησή μας, καθώς και ο Καναδάς. Η θεσμική ασφάλεια της ε, οργάνωσής μας εξασφαλίζεται με ετήσια επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η στήριξη αυτή είναι πολύ σημαντική ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα της CED και υπολογίζουμε και στη δική σας στήριξη. Στη διάρκεια του 2016 η οργάνωσή μας προχώρησε σε πλήρη αξιολόγηση από εξωτερική από εξωτερικούς αξιολογητές Ολλανδούς και αυτοί ε, βρήκαν ότι ήταν σημαντική η δραστηριότητά μας για να χρηματοδοτήσουμε υποχρηματοδοτούμενες δραστηριότητες και φορείς. Η αξιολόγηση αυτή τόνισε επίσης ότι η δραστηριότητα μας αυτή είχε συμπληρωματικό χαρακτήρα για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ταχείες απαντήσεις που επιτρέπουν να επιλέξουμε τους πιο υποσχόμενους φορείς οι οποίοι αξίζουν την χρηματοδοτική μας στήριξη. Στη Μολδαβία, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε στήριξη σε δύο σημαντικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που επέτρεψε να αποφευθεί το κλείσιμό τους στο άμεσο μέλλον. Η τηλεοπτική σταθμή υφίσταντο τρομερή πίεση με ε, έλλειψη διαφημίσεων και με σημαντικό ανταγωνισμό από τους άλλους φορείς. Σε χώρες όπως Αίγυπτος, Ρωσία, Λευκορωσία, Αζερβαϊτζάν, όπου είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες της κοινωνίας των πολιτών, η ΕΕ προσφέρει σημαντική βοήθεια σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Η στήριξη λοιπόν της ΙΕΤ υπήρξε ζωτική σημασία για τα κινήματα αυτά. Στη Συρία η EED έχει στηρίξει τις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών και συνεχίζει να στηρίζει μια πολυφωνική Συρία με υποστήριξη σε τοπικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού και ιδίως σε δύσβατες περιοχές. εκτός από την εργασία εντός της χώρας αυτής, στηρίζει και προσφυγικές κοινότητες σύρων στον Λίβανο για να καταδείξουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε να μειωθεί η προσφυγική πίεση. Εάν μπορέσουμε δηλαδή να βοηθήσουμε τις χώρες όπου κατοικούν οι πρόσφυγες και όπου οι άνθρωποι αυτοί για τόσα πολλά χρόνια έχουν τόσο λίγες δυνατότητες να δράσουν. Η ετήσια έκθεσή μας, την οποία σας έδειξα προηγουμένως και ελπίζω να την έχετε λάβει, σας δίνει και άλλες λεπτομέρειες και παραδείγματα της εργασίας μας. Και βεβαίως θα την βρείτε, όπως είπα, και διαδικτυακά. Περιλαμβάνουμε μάλιστα και φωνές φορέων από επιτόπου δραστηριότητές μας, on the field. Και αυτές οι συνεντεύξεις δείχνουν ποιες είναι οι σημαντικές προσπάθειες που καταβάλουν τα πρόσωπα αυτά και οι θυσίες που κάνουν. Σε μία συνέντευξη είναι η ιστορία του Αμπδεαρχήμ Μάντι από την Τινησία που πέρασε 20 χρόνια στη φυλακή λόγω πολιτικής δραστηριότητας πριν από την Επανάσταση του 2011 και τώρα που η χώρα του η Τινησία βρίσκεται σε δημοκρατική μετάβαση εργάζεται υπέρ της ισότητας των φύλων στη χώρα αυτή. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ε, φορέων που στηρίζουμε δεν επιζητούν την επανάσταση. Θέλουν μια αξιοπρεπή ζωή. Συνήθω πρόκειται για νέου ανθρώπου που έχουν όνειρο, όνειρα για το μέλλον και είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν στην ε, ζωή τη κοινότητα στην οποία ζουν. Στην διάρκεια του περασμένου έτου, όπω είπα και στην αρχή, παρατηρήσαμε σημαντική αλλαγή του εργασιακού μα περιβάλλοντο και εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπιστώνουμε μια σύγκληση για θέματα soft power που όμως γίνονται πλέον τμήματα της hard power ε, ασφάλειας. Συναντήθηκα τον προηγούμενο μήνα με εκπροσώπους της φιλανδικής κυβέρνησης για μια προσπάθεια που αναλαμβάνει το Υπουργείο Άμυνάς τους. Παρόλο που η ED δεν έχει σχέση με, τη, με, με τον παραδοσιακό προβληματισμό ασφάλεια, αντιλαμβάνεται την ανάγκη να δραστηριοποιηθεί και αυτό δεν πρόκειται μόνο με την περίπτωση. Το 2016 διαπιστώσαμε ότι εκεί που στηρίξαμε ε, στρογγυλές τράπεζες για τον τύπο κτλ. αλλάζουν σιγά σιγά όλη την παρουσία των κυβερνητικών δυνάμεων. Πρόκειται για νέο φαινόμενο και νέα φαινόμενα μάλλον και για μια νέα πραγματικότητα η οποία προσφέρει ευκαιρίες αλλά σημαίνει και προκλήσεις και δίνει μεγαλύτερη πολιτική σημασία στο έργο μας. Όλο και περισσότεροι δε πολιτικοί αντιλαμβάνονται την σημασία που έχουν αυτά τα project τα οποία μπορούν να έχουν εκτός από τη soft power διάσταση και μια σκληρή διάσταση. Και υπάρχει μάλιστα κατανόηση ότι τα πιο επιτακτικά θέματα στην σημερινή πολιτική ατζέντα όπως η προκλήση του προσφυγικού, η ριζοσπαστικοποίηση των νέων στην σε Ανατολή και άλλα έχουν άμεση σχέση με την υποστήριξη δημοκρατικά προγράμματα που δίνει η ΕΔΗ καθώς και άλλοι φορείς. Ταυτόχρονα όμως η σύγκληση ασφάλειας και δημοκρατία αποτελεί και μια παγίδα. Ορισμένοι πολιτικοί στην Ευρώπη πάνε να ισορροπήσουν το ένα κατά του άλλου, προωθώντας την ψευδέστηση ότι δήθεν τα πολιταρχικά καθεστώτα μπορούν να προσφέρουν κάποιες ρεαλιστικές λύσεις για την ανάπτυξη. Σε περίοδους κρίσεων οι πολιτικές θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές, ωστόσο πάντα βασισμένες σε αρχές και αξίες. Οι ακτιβιστές που υποστηρίζουν το έργο μας αρχές και αξίες έχουν κρίσιμη σημασία για μας και θα πρέπει να ζητούμε σε αιτήσια βάση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικότερα να υποστηρίζουν την αποστολή της EED και να μην κάνουν συμβασμούς για βραχυπρόθεσμα κέρδη. Μόνο έτσι θα παραμείνουμε αξιόπιστος εταίρος για όλους τους ακτιβιστές που χρειάζονται την δράση και τη συνεργασία μας. Τελειώνω με ένα γενικό σχόλιο μακροπρόθεσμα. Το να παραμείνουμε πιστοί σε αυτές τις δημοκρατικές αξίες και αρχές είναι και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις, την, τα ισχυρά σημεία των κοινωνιών μας. Και αυτά που πράττουμε εμείς και υπέρ των ακτιβιστών στις περιοχές αυτές αντανακλούν θετικά και στις δικές μας κοινωνίες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ευχαριστώ θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας το ΕΛΚ πρώτα, ο κύριος Βέντα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λυπάμαι που άργησα λίγο, αλλά ήμουνα στην Επιτροπή Ανάπτυξης, όπου είχαμε δημόσια ακρόαση για την ερεσιμότητα και την αναπτυξιακή βοήθεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ανταλλαγή αυτή απόψεων που μπορούμε να έχουμε με τον κύριο Πομιανόφσκι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία. Εδώ μιλάμε βέβαια για τις δράσεις εκείνες οι οποίες βεθούν σε καλύτερη συνδυτοποίηση των Ευρωπαίων στην υποστήριξη διαφόρων κινημάτων υπέρ της δημοκρατίας πρέπει να σκεφτούμε τη γειτονιά μας στις χώρες ε, ανατολικά της Ευρώπης, νότια της Ευρώπης, τη Βόρεια δηλαδή. Όντως το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται σίγουρα ευελιξία. Λαμβάνεται υπόψη ένα σωρό παράγοντες. Συνεπώς, πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ εγώ στην στήριξή σας στη Συρία. Έξι χρόνια εμφύλιο πόλεμο έχουμε στη Συρία. Η κατάσταση δυστυχώς επιδεινώνεται αντί να βελτιώνεται. Οπότε η ερώτησή μου είναι, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα, βλέπετε μήπως φως στην άκρη του τούνελ. Οι Σύριοι εμπνέονται από τις Ευρωπαϊκές Αρχές Δημοκρατίας και Πλουραλισμού. Πιστεύετε ότι μπορούμε να τους στηρίξουμε. Είναι κάποιες ομάδες, ε, χρειαζόμαστε κάποιον επικεφαλής κοινωνικών ομάδων. Γιατί όταν κανείς σκέφτεται το μέλλον μιας τέτοιας χώρας που έχει περάσει από πόλεμο, προφανώς και χρειάζεται κάποια ηγετική μορφή. Τι λέτε γι' αυτό. Η κυρία Φωτίγκα τώρα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ε, ευχαριστώ, κύριε Πρέσβη. Συγχαρητήρια για το έργο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Δημοκρατία. Και πέρυσι διαπίστωσα πως αξιόλογο είναι το έργο σας, εξετάζοντας ακριβώς το έργο αυτό εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Έχει να κάνει όχι με την ε, Ρωσική Ομοσπονδία αυτή καθεαυτή, αλλά με τα κατεχόμενα, τα οποία άμεσα ή έμεσα κατέχονται. Πώς μπορούμε να επισημάνουμε τα προβλήματα αυτά. Οι τάρταρες στην Κρυμαία, για παράδειγμα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για αυτούς. Πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε την ύπαρξη κάποιων προγραμμάτων υπέρ αυτών. Οι θέματα ενημέρωσης, βοήθεια προς την κοινωνία. Είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας. Καταλαβαίνω ότι η ερώτησή μου είναι δύσκολη, οπότε και η απάντηση θα είναι δύσκολη, αλλά παρόλα αυτά την κάνω. Και έπειτα στην Αυκαζία, ως αιτία, πώς μπορούμε να επηρεάσουμε στα εδάφη αυτά τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Πρασίνων τώρα, ε, ο κύριος Ρίκ. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Μέσεριξ, για την παρουσία σας εδώ. Δεν θα χρονοτριβήσω με ευχαριστίες. Ξέρουμε ότι το έργο σας είναι πολύ σημαντικό και το ταμείο σας επίσης. Οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένο. Αλλά έχω δύο κάπως πρακτικές ερωτήσεις. Έχουν να κάνουν όμως και με τη γενική πολιτική σας. Το πρώτο είναι το εξή. Το τελευταίο χρόνο, μισή χρόνο, οι δραστηριότητες σας έχουν επεκταθεί γεωγραφικά. Οι δωρητέ πρέπει να ξέρουν τι εξελίξεις υπάρχουν επιτόπου, κατά πόσο ε, ανταποκρίνονται σε αιτήματα που έρχονται από συγκεκριμένες περιοχές ή όχι. Οπότε, πώς το λύνεται αυτό. Εσείς επικεντρώνεστε περισσότερο στην ε, Μολδαβία και την Αρμενία επειδή ε, πιεστήκατε εκ των έσω ή επειδή σας το ζήτησαν οι χώρες αυτές. Και δεύτερον, για τις επιχορηγήσεις που δίνονται και αυτοί που τις δίνουν. Έχετε επαφές με αυτούς που δίνουν τις επιχορηγήσεις ε, τακτικά, μόνιμα, πώς. Ο κύριος Σαφάζε τώρα από το ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο μένα με εκπλήσει και χαίρομαι που η χώρα μου η Γαλλία δεν συμμετέχει. Αυτό που με εκπλήσει λοιπόν είναι η αλαζονία στην προπαγάνδα. Το ότι κεντρικά ε, οργανώνεται η προπαγάνδα αυτή όπως κάνετε εσείς. Κοίταξα κάποια σημεία Ουκρανία, Μαϊντάν. Εσείς φτιάχνετε την ιστορία. Δεν λέτε πώς έγιναν τα πράγματα. Συρία. Πώς μπορείτε να ξεχάσετε την στήριξη προς τις τρομοκρατικές ομάδες από κάποιες δημοκρατικές χώρες ή ακόμα από τις δικές μας υπηρεσίες πληροφοριών που φάνηκε αυτό. Η χώρα μου για παράδειγμα. Ερχόσαστε εδώ με τα γνωστά στερεότυπα. Ε, φέρνετε εδώ την θεωρία των ειδών. Εγώ αμφισβητώ μια τέτοια θεωρία και δεν την αμφισβητούμε μόνο εμείς που πιστεύουμε, αλλά εσείς δεν τηρείτε καν την ελευθερία στη θρησκεία. Παραπληροφορείτε και λέτε ότι αυτό αποτελεί εργαλείο για την ε, πληροφόρηση και για τη δημοκρατία. Εγώ συμμετείχα μαζί με άλλους στην αντιπολίτευση για να πέσει το τείχος του Βερολίνου. Ε, και τώρα το ίδιο πρέπει να κάνω. Όπως έκανα παλιά κατά του κομμουνισμού, τώρα πρέπει να κάνω το ίδιο κατά του συστήματος που εσεί εκπροσωπείτε, που είναι ένα σύστημα προπαγάνδας, ανυπόφορο. Ευτυχώ ξυπνούν οι λαοί και δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε όπω κάνατε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι μιλητέ μα. Θα σα δώσω ένα τετράλεπτο να συνοψίσετε. you Thank you Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις άκρος θετικές απόψεις εκτός μίας, της τελευταίας. Θα ξεκινήσω από τη μειοψηφία. Η Γαλλία στηρίζει το Ταμείο. Δεν συνεισφέρει ακόμα, αλλά είναι συνεισφορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω αυτού του μηχανισμού μας υποστηρίζει. Και βρίσκεται και στο διοικητικό μας συμβούλιο. Συμμετέχει στις συζητήσεις, σχεδιάζει τις αποστολές μας, καθορίζει προτεραιότητες, βασικές προτεραιότητες. Πρόσφατα, πριν από μια εβδομάδα, επεσκέφθη το Παρίσι και είχαμε στο κέντρο ΕΣΤΕΠΟ εξωτερικών είχαμε συζητήσει για το θέμα αυτό και ε, ήταν θετικές οι απόψεις που άκουσα πλευράς Γαλλίας. Θέλω να πω ότι ακούω τις απόψεις της γαλλικής κυβερνήσεως όσον αφορά τις θέσεις της χώρας εν Άκουσα όμως τα σχόλιά σας. Με τα περισσότερα σχόλιά σας διαφωνώ. Όσον αφορά τη Συρία, ο Σβέντα έθεσε ένα ερώτημα Θέλουμε να αυξήσουμε στο μέτω του δυνατού την υποστήριξη στους ανθρώπους που ζουν στους καταβλισμούς προσφύγων. Έχουμε εκατομμύρια σύρων οι οποίοι δεν προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη, είναι κοντά στην πατρίδα τους και ονειρεύονται να επιστρέψουν όποτε μπορέσουν. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εκεί για μια μελλοντική νέα Συρία έχουν μείνει μόνοι τους. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα ε, για την αγωγή του πολίτου, για την παιδεία, κυρίως για την εκπαίδευση των νέων. Ξέφυγαν ένα δεκαετής σήμερα, πριν από έξι χρόνια, ξέφυγε τη Συρία. Τα έξι χρόνια ζει σε καταπλησμούς προσφύγων. Αυτό το παιδί, α, έφυγε 12, τώρα είναι 18. Διακόπηκε η εκπαίδευσή του. Ποιος θα προσλάβει αυτό το παιδί. Ποιος θα προσπαθήσει να στατολογήσει αυτό το παιδί. Έναντι ποιον είναι πιο ευάλωτος. Πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία, τα κατάλληλα μέσα που πρέπει να ξεπερνούν το Ευρωπαϊκό Τάμιο για τη Δημοκρατία. Μπορούμε να δρομολογήσουμε κάποια προγράμματα, έχουν περιορισμένους πόρους, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο απόθεμα που έχουμε για μελλοντική λύση και πρέπει να επενδύσουμε πολλά εκεί. Ευχαριστώ κυρία Φωτίγκα για την υποστήριξή σας. Χρήσιμα αυτά που είπατε. Όπως είπατε, συνεργαζόμαστε σε πολλούς τομείς. Με τη συγκεκριμένη ερώτησή σας τώρα. Για τους Τατάρους της Κρυμαίας. Συνεργαζόμαστε μαζί τους μέσω προγραμμάτων εντός Κρυμαίας και εκτός αυτής. Εδώ το Ταμείο ειδικεύεται να κινείται σε εχθρικά περιβάλλοντα δεν μπορούμε να δημοσιοποιούμε τα στοιχεία της, ε, του προγράμματος αυτού μόνο και μόνο για λόγους ασφαλείας του προσωπικού. Όσον αφορά την επέκταση, ο Τάμας Μοίρας, το νέο μέλος, ζήτησε για τη γεωγραφική επέκταση. Αυτό απαιτεί περισσότερα χρήματα, προφανώς. Έχουμε επεκτείνει τη γεωγραφική μας κάλυψη. Δυστυχώς όχι συμφωνά ανάλογα με την ε, αύξηση του προπολογισμού. Αυξάνεται ο προπολογισμό μας, αλλά με μικρότερους ρυθμούς από τη η γεωγραφική μας ε, επέκταση. Άρα δεν έχουμε ταχύτητα πορείας ε, στις νέες περιοχές. Αναλύουμε τις ανάγκες τώρα και ανταποκρινόμεθα σε αρχικές αιτήσει. Όμως έχουμε ακόμα παραδείγματα προγραμμάτων που προωθούνται σε νέες περιοχές, με μία εξαίρεση. Από δύο πήραμε περισσότερα χρήματα για την ε, Ευρασία και μπορέσαμε να κινηθούμε ταχύτερα. Και μας βοήθησε η συμπληρωματική χρηματοδότηση να κινηθούμε έτσι. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Αν έχετε κι άλλες, με τα χαράς να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που δώσατε. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Δεν έφτασαν ακόμα οι φιλοξενούμενοι μας. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το επόμενο σημείο θα συζητηθεί και κλεισμένο των θυρών. Μόνο μέλη και προσωπικό πολιτικών ομάδων και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να είναι παρόντες. Οπότε παρακαλώ να αποχωρήσουν από την αίθουσα εκείνοι που δεν δικαιούνται να παρίστανται στις συνεδρίες και κλεισμένο των θυρών.